Good morning, ladies and gentlemen. Um, we're about to start. It's Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 9 και 5. Ας ξεκινήσουμε διότι έχουμε πολλές αναφορές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το μόνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι το σημείο 26 είναι η αναφορά 0188 κάθετος 2015 της Βουλγαρίας. Θα συζητηθεί σήμερα πριν το 25, διότι πρέπει να αποχωρήσει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής στις 10.30. Αν συμφωνείτε λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία διαφωνία, οπότε ξεκινάμε. Η πρώτη μας αναφορά είναι η παριθμόν 750-2015 Ολλανδού αναφέροντος. Δεν είναι παρόν. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως έχει στείλει ένα επιπλέον έγγραφο με τέσσερις ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, ε, στάλει στις 29 Ιουνίου. Ε, και θα μας παρακολουθεί από το διαδίκτυο. Δεν είναι παρόν ο αναφέρον. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο αναφέρον ε, και στην ε, αναφορά και στο έγγραφο που λάβαμε εκ των υστέρων ε, θίγει τρία βασικά θέματα. Ζητά να εστιαστούμε επιπλέον στην μείωση των εκπομπών διευσυδίου του άνθρακα στην οδηγία για την απόδοση των κτηρίων Επίσης ε, ζητά διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών ε, και κατά τον υπολογισμό της ε, κατανάλωσης ενέργειας καθώς και και φύγει επίσης την προσέγγιση στις κάτω χώρες όσον αφορά την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Σε απάντηση λοιπόν αυτών των ε, τριών ζητημάτων πρέπει να αναφέρουμε ότι οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων επικεντρώνεται κυρίως στην ενεργειακή απόδοση. Αυτό ήταν ε, η επιλογή του συνομοθέτη, κάτι όμως που έχει και θετικές επιπτώσεις ε, στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ο νομοθέτης επέλεξε να αφήσει σε εθνικό επίπεδο τα προγράμματα για την ε, σήμανση. Είναι όμως ε, σημαντικό να αναφέρουμε ότι παρόλα αυτά η οδηγία αναφέρει ρητά την ε, δυνατότητα να να γίνουν αυτά που ζητάει ο αναφέρον, ε, για παράδειγμα η ε, διαφοροποίηση ανάμεσα στα, στις κατοικίες ε, και σε άλλα κτίρια όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά τον τρόπο μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας, το να γίνεται αιτησίως. Δηλαδή και αυτό είναι μια δυνατότητα που αναφέρεται στην οδηγία. Επίσης σημαντικό ε, είναι να αναφέρουμε ότι η οδηγία αναφέρει και ενεργειακή απόδοση και ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να ισχυριστούμε ότι η οδηγία αυτή εμποδίζει την βιώσιμη κατανάλωση ενέργειας, αντιθέτως την προωθεί. Επίσης, όσον αφορά την προτιμητέα προσέγγιση, Η προσέγγιση αυτή αποτελεί επιλογή του εθνικού νομοθέτη με βάση τις δυνατότητες που προβλέπονται στην οδηγία. Υπάρχει ευρύ περιθώριο ευελιξίας στην οδηγία. Σημαντικό όμως είναι να αναφέρουμε επίσης ότι αναθεωρείται αυτή τη στιγμή η οδηγία με στόχο υιοθέτησης πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχές Οκτωβρίου μάλλον. Δεν έχει ληφθεί απόφαση ακόμα όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας, άρα δεν μπορούμε ακόμα να σας πούμε τι μορφή θα έχει η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανείς που θέλει να πάρει το λόγο. Από ό,τι βλέπω όχι. Αναμένουμε την αναθεώρηση που είπατε, το φθινόπωρο από ό,τι καταλαβαίνω. Προτείνω λοιπόν να παραμείνει σε κρεμότητα η αναφορά αυτή ώστε να μπορέσουμε να ενημερωθούμε καλύτερα σχετικά με το τι συμβαίνει. Αφήνουμε λοιπόν ανοιχτή την ε, αναφορά αυτή. Um, we should be doing another petition, petition number θα έπρεπε να προχωρήσουμε στην αναφορά υπαριθμών 22, αλλά με ενημερώνουν ότι δεν είναι ακόμα παρόν ο εκπρόσωπο ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να προχωρήσουμε λοιπόν στην ε, αναφορά 23 και θα περάσουμε στην 22 όταν καταφτάσει ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή, διότι ούτε και ο αναφέρον είναι παρόν. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο 23, αναφορά 0496 του 2015 αναφέροντος βρετανική Ιθαγένειας ε, και πάλι δεν είναι παρόν ο αναφέρον. Ε, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η αναφορά αναφέρεται στην εξής κατάσταση. Ε, Βρετανός επίκος δεν λαμβάνει πια ηλεκτρικό ρεύμα και αέριο ε, τα ελάμβανε στο παρελθόν ε, μέσω μιας ε, σύμβασης που υπογράφουν οι εταιρείε κατασκευής των κτηρίων με τις εταιρείε. Κατόπιν ο αναφέρον ζήτησε ένα κανονικό εγχώριο συμβόλαιο με τον πάροχο ενέργειας. Ωστόσο, η εταιρεία παροχή ενέργεια χρειαζόταν πιστοποιητικά ότι έχει κατασκευαστεί σωστά το κτίριο και ότι είναι κατάλληλο ω ανθρώπινη κατοικία. Εξετάσαμε προσεκτικά την αναφορά και συνομιλήσαμε με ε, την ε, Ισπανική Ρυθμιστική ε, Αρχή για την Ενέργεια, η οποία αναγνώρισε το πρόβλημα. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι στην νομοθεσία που να εμποδίζει την παροχή ενέργειας στον αναφέροντα. Το πρόβλημα ήταν η έλλειψη των κατάλληλων πιστοποιητικών. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεραίνει με λύπη και καταλαβαίνοντα το πρόβλημα του Βρετανού Επικοού ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το πρόσωπο αυτό, διότι το πρόβλημα οφείλεται στην έλλειψη των κατάλληλων πιστοποιητικών. Τον συμβουλεύουμε λοιπόν να έρθει σε επαφή με τις ε, περιφερειακές και τοπικές αρχές που έχουν να κάνουν με την ε, καταχώρηση των κτηρίων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνω, το θέμα αυτό πια ε, αφορά εθνικές αρμοδιότητες. Και από ό,τι μας είπατε, δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να κάνουμε. Όχι δυστυχώς, λέει ο μιλητής. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να κάνουμε. Ένα ευρωβουλευτή όμως θέλει πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση. Είναι αδύνατον να λάβει το πιστοποιητικό αυτό αναφέρον. Είναι κάτι εύκολο. Διότι το πρόβλημα είναι το πιστοποιητικό από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ήθελα να γνωρίζω. Είναι ε, απλή περιέργεια, πολιτική περιέργεια βέβαια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Δεν είναι αδύνατον να λάβει το πιστοποιητικό αυτό ο αναφέρον. Δυστυχώς όμως από τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να κάνουμε. Μελετήσαμε την αναφορά και φαίνεται ότι για να καταχωρήσει κανείς ε, την κατοικία του πρέπει να έχει πιστοποιητικό ότι είναι κατάλληλο ως κατοικία. Είναι λοιπόν κάτι που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο αναφέρον με τις τοπικές αρχές. Εμείς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να διευκολύνουμε τη διαδικασία, διότι αφορά τη σχέση του προσώπου αυτού και των τοπικών αρχών. Ε, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά έκανε αίτηση να λάβει το πιστοποιητικό αυτό, διότι εάν έχει υποβάλει αίτηση και δεν το έλαβε, τότε υπάρχει πρόβλημα. Εάν απλά δεν έκανε την αίτηση, τότε είναι άλλο θέμα. Από την αναφορά φαίνεται ότι είχε υποβάλει αίτηση για να λάβει το πιστοποιητικό και περίμενε να το παραλάβει αναγνωρίζει δηλαδή την ε, διαδικασία αυτή, αλλά στο μεταξύ έχει διακοπεί η παροχή ε, ηλεκτρικού και αερίου και αυτό είναι το πρόβλημα. Πρόεδρος, ε, από ό,τι καταλαβαίνουμε έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες και ίσως οι ισπανικές αρχές δεν είναι ακόμα ικανοποιημένες όσον αφορά την έκδοση του πιστοποιητικού. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε τέτοια θέματα και με όλη την καλή διάθεση που έχουμε να βοηθήσουμε δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώ, ε, λοιπόν ε, νομίζω πρέπει να προτείνω να κλείσει η αναφορά αυτή. Υπάρχουν παρατηρήσει σχετικά με αυτό. Ωραία, θα ενημερώσουμε τον αναφέροντα ότι κλείνει η υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. We're moving on now to petition. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 24, αναφορά 0529-2014, Ιταλική Ιθαγένειας και πάλι ο αναφέρον δεν βρίσκεται εδώ. Παρακαλώ το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε λάβει αυτή την αναφορά μόλις την περασμένη εβδομάδα δυστυχώς. Επομένως ε, δεν μπορώ να σας δώσω μια πλήρη και οριστική εκτίμηση, μη κάποιες προκατακτικές απόψεις μόνο. Ο αναφέρον καταγγέλει ότι για μια περίοδο τριών ετών, για το 2014 στάλει η αναφορά, δεν έχουν υπάρξει κατάλληλες μετρήσεις από το 2011. Επίσης, ο αναφέρον έχει βάλει φωτοβολταϊκά στη στέγη και ισχυρίζεται ότι η παραγωγή αυτή δεν έχει ληφθεί υπόψη στο τελικό του τιμολόγιο. Γιατί ακριβώς δεν γίνονταν σωστά η τιμολόγηση. Ο αναφέρον λοιπόν καταγγέλει ότι δεν έχει λάβει διαφανείς πληροφορίες, ότι η παραγωγή ηλιακή ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά του δεν ε, συνυπολογίζεται στο τελικό τιμολόγιο. Από πλευρά Επιτροπή, σε πρώτη ανάλυση μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση που περιγράφει ο αναφέρον συνδέεται ρητός με τις υποχρεώσεις ε, των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών μελών υπό την οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια και την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση να παρέχουν τιμολόγια και σχετικές πληροφορίες βάσει ακριβών μετρήσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ένα έτος. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα προετοιμάσουμε πλήρη γραπτή απάντηση εντός των επόμενων εβδομάδων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Με βάση τις περιστάσεις θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά λοιπόν γιατί δεν είχατε και εσείς προφανώς και το χρόνο να ενημερωθείτε πλήρως. Δεν έχουμε άλλη επιλογή λοιπόν από το να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Δεν ξέρω τα μέλη θα ήθελα να πάρουν το λόγο ως προς αυτή την αναφορά. Όχι. Εντάξει, μένει ανοιχτή η αναφορά αυτή λοιπόν. Ευχαριστώ. Σημείο 26. Αναφορά 188 του 2015 από αναφέρονται βουλγαρικής ηθαγένειας. Και πάλι δεν είναι εδώ αναφέρον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν. Good morning, thank you. Καλημέρα, ευχαριστώ. Αυτή η αναφορά αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή και τον ε, ε, τον ε, κλάδο παραγωγής ενέργειας. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι ο αναφέρον αρχικά θέτει ένα ζήτημα ορολογίας που αφορά τι, τι νέες τροπολογίες ε, στην βουλγαρική νομοθεσία σε ό,τι αφορά την πώληση και τη διανομή. Εξετάσαμε την νομοθεσία και δεν έχουμε βρει κάτι στην ενεργική νομοθεσία που να ρυθμίζει ακριβώς πώς θα πρέπει να ορίζεται ε, η διανομή της θέρμανσης. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι λοιπόν προς αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι γενικότερου χαρακτήρα και για τον τρόπο οργάνωσης της αγοράς θέρμανσης. Ο αναφέρον ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δραστηριοτήτων της παραγωγής ενέργειας, της μεταφοράς και διανομής της. Και πάλι υπάρχει η ρύθμιση σε αυτό το τομέα για ε, την ηλεκτρική ενέργεια και για το φυσικό αέριο, αλλά όχι για τη θέρμανση. Επομένω, δεν υπάρχει κάτι στην βουλγαρική νομοθεσία που να αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκαιο. Μετά, έχετε ζήτημα για το πώ ε, προσδιορίζονται οι όροι και προποθέσει για τι συμβάσει ε, αυτή τη οικιακή θέρμανση. Αυτή τη στιγμή είναι οι πάροχοι που καταρτίζουν αυτού του όρου και μετά εγκρίνονται από τι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ. Και πάλι δεν υπάρχει κάτι στις οδηγίες περί αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας που να ορίζει πώς ακριβώς θα εγκρίνονται αυτοί οι όροι από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή για τη θέρμανση. και μελετήσαμε σε μεγαλύτερο βάθος ε, την υπόθεση στο πλαίσιο των προϋποθέσεων της οδηγίας ενεργειακής απόδοσης για τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, ιδίως κατά πόσο η τιμολόγηση ε, ήταν αναλογική. Και διαπιστώσαμε ότι αυτός ο μηχανισμός με την έγκριση από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή όντως δύναται να διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Επομένω και εδώ δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει κάτι. Το τελευταίο σημείο το αναφέροντα είναι για μια αποτεθέμενη άδικη ε, μορφή αυτών των όρων και προποθέσεων και για την αδυναμία των ε, βούλγαρων υπηκόων να καταγγείλουν αυτούς τους ε, όρους και προποθέσεις. αλλά θεωρούμε, από όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, ότι οι Βούλγαροι υπήκοοι διατηρούν τη δυνατότητα να ε, απευθυνθούν στα αστικά δικαστήρια σε ό,τι αφορά ε, τα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειάς τους και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα για τους Βούλγαρους υπηκόους και τους παροτρύνουμε να έρθουν και σε επαφή με την Επιτροπή για την Προστασία του Καταναλωτή. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τα μέλη έχουν το λόγο. Παρακαλώ κύριο Βαλέσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την αρχή της επικουρικότητας. Και ο αναφέρον θεωρώ ότι θα πρέπει να απευθυνθεί στις ε, εθνικές αρχές και στα αστικά δικαστηρία της Βουλγαρίας. Δεν βλέπω τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Προτείνω να κλείσει η αναφορά αυτή. Κάτι άλλο. Συμφωνώ λέει ο κύριος Άμπρας. Ευχαριστούμε. Και εγώ συμφωνώ, λέει η Πρόεδρος. Από ό,τι βλέπουμε είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Οι εθνικές αρχές πρέπει να το αναλάβουν. Προτείνω λοιπόν να κλείσει αυτή η αναφορά. May I take you now to item 22, the representative of the Λοιπόν, για το σημείο 22 τώρα θα επιστρέψουμε, γιατί ήρθε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε λοιπόν στην 2547 του 2013. Ο αναφέρον δεν είναι εδώ και πάλι. Όμως με ενημερώνουν ότι μέσω διαδικτύου θα μας ε, παρακολουθεί, θα παρακολουθεί τη συζήτηση. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, αυτή η αναφορά σχετίζεται με τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία το 2013. Οι καταναλωτές λοιπόν χαμηλής κατανάλωσης έρχονται αντιμέτωποι με αύξηση 40% στα τιμολογιά τους. Η θέση της Επιτροπής προς αυτό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ιδίως το τρίτο ενεργειακό πακέτο, ε, παρέχει ε, ευρύ περιθώριο ευελιξίας για τις εθνικές αρχές να προσδιορίσουν ε, τις τιμές. Ωστόσο, η οδηγία ενεργειακής απόδοσης προβλέπουν κανόνες με τους οποίους οι τιμές των δικτύων, οι χρεώσεις των δικτύων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και ορισμένα στοιχεία ενεργειακής απόδοσης και σταθερότητας. Μέχρι το 2013 το σορευτικό έλλειμμα ήταν 30 δις ευρώ. Επομένως, κρίθηκε απαραίτητη μια μεταρρύθμιση της αγοράς. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, χαιρέτησε αυτή τη μεταρρύθμιση. Ήταν απαραίτητο λοιπόν να περιοριστούν οι επιδοτήσεις για κάποιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα ε, σταθερά στοιχεία των τιμολογίων έπρεπε να απελευθερωθούν. Και αυτό δείξει στην αύξηση των τιμών που αναφέρεται και στην αναφορά. Από τότε οι ευρωπαϊκές ε, πρωτοβουλίες πολιτικής για τον ε, ενεργειακό κλάδο παρέχουν ένα πλαίσιο συζήτησης ως προς ε, την πρωτοβουλία αυτή πολιτικής και σύμφωνα με την σημερινή θέση οι εθνικές αρχές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για τον προσδιορισμό των ε, τιμών και χρεώσεων για μία ε, αναλογική κατανομή θα πρέπει όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Contributions from the floor. Τα μέλη έχουν το λόγο παρακαλώ για αυτή την αναφορά. Yes. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι κέριο ζήτημα. Για όλους. Και είναι σαφές ότι στην Ισπανία η ενέργεια είναι απίστευτα ακριβή. Με τις πιο υψηλές τιμές στην Ευρώπη. Και αυτό το 40% είναι προβληματικό, πιστεύω. Από ό,τι βλέπω ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι απόλυτα σίγουρη ποια πρέπει να είναι η θέση της. Προτιμώ λοιπόν να διερευνήσουμε περαιτέρω την υπόθεση, να το συζητήσουμε κι άλλο και στη συνέχεια να αποφασίσουμε πιο μετά. Προτείνω λοιπόν να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Συμφωνώ. Από ό,τι βλέπω η Επιτροπή ακόμα εξετάζει την υπόθεση, οπότε να την αφήσουμε ανοιχτή. Τι ωραία που συμφωνούμε όλοι. Σήμερα το πρωί τουλάχιστον. Ωραία, συμφωνώ, δεν υπάρχουν επαρκεί πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μείνει ανοιχτή η αναφορά λοιπόν μέχρι που να έχουμε τα στοιχεία για να λάβουμε μια απόφαση. Why? Because the previous point is not yet ready. It's 25. Yeah, so there is. I am informed that we will have to jump. Ε, το 25 θα το αφήσουμε προς το παρόν. Πάμε στο 27. Για τεχνικούς λόγους. 0281 του 2011 από αναφέροντα βουλγαρικής ηθαγένειας και πάλι δεν είναι εδώ ο αναφέρον, το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συνοψίσω το υπόβαθρο της αναφοράς, γιατί καταχωρήθηκε το 2011. Έχουν περάσει λοιπόν αρκετά χρόνια. Αρχικά η αναφορά αφορούσε για τη μη μεταφορά της ε, τρίτης δέσμης ε, για την ενέργεια. Το 2013 όμως όταν μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία, στην βουλγαρική νομοθεσία ε, η δέσμη αυτή, ο αναφέρον έδωσε περαιτέρω στοιχεία για την υποτιθέμενη παράβαση του κοινοτικού δικαίου από την βουλγαρική νομοθεσία. Και η Επιτροπή έχει ήδη ενημερώσει το Κοινοβούλιο και τον αναφέροντα στις αρχές του 2014. Από τότε ε, κάνουμε αναλύσει συμμόρφωση με το τρίτο ενεργειακό πακέτο, οι οποίε ολοκληρώθηκαν ε, στα τέλη της περασμένη χρονιάς. Προετοιμάζουμε την τελική μα ε, γνώμη για να απαντήσουμε με οριστικό τρόπο και στον αναφέροντα σύντομα. Όμω τώρα θα ήθελα να στραφώ στο περιεχόμενο τη αναφορά. Ο αναφέρον έθιξε τρία ζητήματα. Το πρώτο ήταν ότι οι καταναλωτέ ηλεκτρική ενέργεια δεν έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια με διαφανή τιμέ στη Βουλγαρία. Το δεύτερο ήταν ότι δεν υπήρχαν κανόνες που να έχουν εισαχθεί στην Εθνική Νομοθεσία τη Βουλγαρίας, ούτω ώστε να υπάρχει πραγματική ε, δικαστική αναθεώρηση ε, στις αποφάσεις της εθνική Ρυθμιστική Αρχής. Και το τρίτο ήταν ότι ε, δεν, μπορούν, δεν μπορούσε να φέρουν να επιλέξει ελεύθερα τον πάροχό του, να αλλάξει δηλαδή πάροχο. Για το πρώτο, για τη διαφάνεια των τιμών. Αυτό αφορά το άρθρο 3 της Οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια. Ε, που αναφέρεται στην διαφάνεια των ε, ενοχικών στις συμβάσεις δηλαδή. Όπως ξέρετε στη Βουλγαρία ακόμα υπάρχουν ρυθμισμένε τιμέ, το οποίο δημιουργεί σημαντικά ε, προβλήματα ελλημάτων στι χρεώσει, γιατί πολλέ φορέ ορίζονται τιμέ κάτω του κόστου. Επομένως πρώτα θα πρέπει να συνεργαστούμε ω Επιτροπή με τι βουλγαρικές αρχέ για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και οι τιμές να καθορίζονται με όρους αγοράς. Το Βουλγαρικό Υπουργείο Ενέργειας το Μάιο φέτος ανακοίνωσε ότι θα απελευθερωθούν οι τιμές και ο μηχανισμός για τον προσδιορισμό των τιμών για τα νοικοκυριά το 2021. Παράλληλα ε, θα ισχύσουν και οι προβλέψεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Ελπίζουμε έτσι να απαντούμε ικανοποιητικά στον αναφέροντα και ελπίζουμε τις τελικές μας απόψεις ε, να τις ε, δώσουμε αρκετά σύντομα. Για το δεύτερο ζήτημα, ε, οι αρχές μας έχουν αναλύσει την βουλγαρική ε, νομοθεσία σε σχέση με την τρίτη ενεργειακή δέσμη και δεν εντόπισαν παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου γιατί Αναφέρει ο ότι δεν υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας, δικαστικού ελέγχου δηλαδή, γιατί το δικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την απόφαση της Εθνικής Ρυθμιστική αρχή. Όμως η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν λέει ότι θα πρέπει το Εθνικό Δικαστήριο να έχει αυτή τη δυνατότητα αναστολή τη άλλη απόφαση. Δεν υπάρχει λοιπόν παράβαση εδώ του κοινοτικού δικαίου. Τώρα που έχει γίνει αυτή η ανάλυση θα ενημερώσουμε σύντομα για τον αναφέροντα. Και για το τελευταίο ζήτημα, το δικαίωμα επιλογής παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, το θέμα ήταν ότι υπήρχε νομική δυνατότητα, αλλά όχι πρακτική. Δεν υπήρχαν τυποποιημένα προφίλ των παρόχων, που είναι μια τεχνική προπόθεση. Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στη Βουλγαρία ε, δημοσιοποίησε αυτά τα προφίλ φέτος πριν από μερικού μήνε και ελπίζουμε να ε, ενημερώσουμε με τι κατάλληλε απαντήσει και τον αναφέροντα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Θέλει κανεί να πάρει το λόγο για αυτό το θέμα. Παρακαλώ, κύριε κουνάμα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι κάτω από το κόστος ηλεκτροενέργειας στη Βουλγαρία αφού η ζωή εκεί θεωρείται χαμηλότερο, ότι έχει χαμηλότερο κόστος. Εγώ ζω στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία και στο Βέλγιο, σε τέσσερι χώρε ταυτόχρονα. Οι πιο, ε, οι πιο δύσκολοι λογαριασμοί έρχονται από τη Βουλγαρία. Η τέρμανση και το ρεύμα σε ένα άνθρωπο, να πούμε μια κατηγητρία, οι μήνε από το Οκτώβριο και μετά έω και το Μάη, δεν αρκεί το μισθό τη να καλύψει τα έξοδα για τέρμανση και ρεύμα στη Βουλγαρία. Ολόκληρο μισθό μιλάμε. Αν δεν δουλεύουν και οι δύο μέλη τη οικογένεια, αποκλείεται να καταφέρει τους μήνες αυτούς, δηλαδή μισό χρόνο δεν έχουν τι να φάνε, δεν έχουν πώ να επιβιώσουν αυτέ τι οικογένειε. Δεν ξέρω πώ είναι χαμηλότερο το κόστο στη Βουλγαρία. Εμένα μου έρχονται πιο μικρές πιο μικροί λογαριασμοί από τη Γαλλία και από την Ελλάδα όσο στη Βουλγαρία, αν ζούμε εκεί τους μήνες αυτούς. Και νομίζω ότι πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να κοιτάξουμε την κατάσταση της Βουλγαρίας με την τοποφικάτσια, με την τέρμαση και με το ρεύμα, γιατί τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε εννιά αυτοκτονίες, οι οποίες είναι με πώς λέγεται, αυτοπυρπόληση και είναι με δήλωση γιατί δεν, μπορούν να πληρώσουν τα, οι λογαριασμοί τους για το ρεύμα και τη τέρμανση. Και ένα άλλο ακόμα το οποίο βγαίνει στο τύπο τελευταία πολύ συχνά, ότι έχουν ξεκινήσει αυτές οι εταιρείε να μην ειδοποιούν τους πελάτες τους, να υπάρχει ένα λογαριασμό έναντι το οποίο το πληρώνουν οι πελάτες και μετά όταν έρχεται ανακυρούς ολοκληρωμένο το λογαριασμό το οποίο δεν φτάνει στο πελάτη, δεν ξέρει ότι πρέπει να πάει να το πληρώσει, ξεκινάνε δικαστήρια και από ένα λογαριασμό το πρέπει να, πρέπει να πληρώσει 300-400 ευρώ, το έρχεται απόφαση δικαστηρίου για 4.000 λέβα. Αυτό είναι πάρα πολλά λεφτά. Γιατί ένα συνταξιούχος του Βουλγαρία παίρνει 60 ευρώ, 70 ευρώ 100 ευρώ το πολύ είναι η σύνταξή του. Ένα μισθό είναι 160 ευρώ. Και πώς να πληρώσω τόσο λεφτά. Από να πάρει τα 200 ευρώ μόνο για να ολοκληρώσει την εποχή. Νομίζω ότι θέλει πολύ καλύτερη μελέτη. Νομίζω ότι αυτές οι τιμές στη Βουλγαρία είναι πολύ ψηλές. Η μίστη είναι πολύ χαμηλή. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Kuneva. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κουνέβα. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Βεβαίως είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τους πάντες. Αν τώρα είναι δική μας αρμοδιότητα να εξετάσουμε τις τιμές, είναι κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι έχουμε επαρκείς πληροφορίες αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από ό,τι βλέπω ακόμα και η Επιτροπή περιμένει περαιτέρω στοιχεία. Προτείνω λοιπόν αυτή η αναφορά να μην ανοιχτεί. Yes, we're also waiting for the finalized... Uh, Περιμένουμε και την οριστική απάντηση της Επιτροπής έτσι κι Οπότε ναι, θα παραμείνει ανοιχτή. Εντάξει. Right, it's a, it's a bit of a backwards and forwards day. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στο σημείο 25. Και πάλι από επικούς βουλγαρικής ηθαγένειας. Έχουμε αρκετέ εδώ. Θα πω τους αριθμούς τους μόνο. Όλοι από τη Βουλγαρία. Οι αναφέροντες δεν είναι εδώ. Όμως έχουμε βίντεο. Τώρα θα δούμε την 892 του 2008. 1542 του 2009, 38 του 2013 και εδώ θα προβληθεί το βίντεο του αναφέροντα τη 256 του 2013 269 του 2013, 2178 του 2013, 0556 του 2014 και 0568 του 2014. Πρώτα όμως Έχουμε βίντεο του κυρίου Ντόνσον Ντούντεφ για τη 038 του 13. Παρακαλώ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, πάνω από τρία χρόνια έχουν περάσει από τότε που υποβάλαμε την αναφορά και πάνω από ένα έτος από τις από τις προσθήκες που λάβαμε στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2015. Στο μεταξύ, η Οδηγία 2011-83 τέθηκε σε ισχύ αφού μεταφέρθηκε στο, στη βουλγαρική νομοθεσία. Εξετάσαμε την, ε, τις παρατηρήσεις της Επιτροπής ε, Αναφορών και έχουμε την εντύπωση ότι δεν έχει καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόβλημα με την ε, εταιρεία το Πλοφικάτσια Σόφια. Έχουμε να κάνουμε με λογαριασμούς ε, συνδρομής και Όταν κάποιος ε, έχει ε, ένα διαμέρισμα, δεν έχει πάντα προσωπικό λογαριασμό. Οι βουλγαρικές αρχές παρακάμπτουν τις διατάξεις της Οδηγίας 2011 κάθετος 83. Διότι εκδίδουν λογαριασμούς ε, όχι σε άτομα, αλλά ε, στο, στην διαχειριστική εταιρεία. Και το δήλωσαν αυτό απέναντι στη Γενική Διεύθυνση για την ε, Ενέργεια. Η εταιρεία διανομής συνάπτει σύμβαση για την διανομή. Η κατάσταση πρέπει να αλλάξει επιγόντως, ε, αλλά οι εταιρείε αρνούνται να εκδώσουν ε, τιμολόγια στο όνομα του πελάτη και σύμφωνα με τους κανόνες για το ΦΠΑ είναι υποχρεωτική η έκδοση τιμολογίου. Πρόκειται για μια μοναδική περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι πουλά ενέργεια στην ε, Ένωση Διοκτητών και έτσι εκδίδονται απλά κοινοποιήσεις προς ε, τους ε, επιμέρους ιδιοκτήτες που δεν έχουν όμως καμία νομική ισχύ. Και αυτές οι μηνιαίες κοινοποιήσεις δεν αντικατοπτρίζουν την ε, πραγματική κατανάλωση. Το κόστος θέρμανσης και ζεστού νερού κατανέμεται στους ε, συνειδιοκτήτες με τρόπο αυθαίρετο. Οι αρχές το γνωρίζουν αυτό εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την πλευρά τους. 250.000 ε, οικογένειες από τη Βουλγαρία ε, έχουν δικαστικές υποθέσεις εις βάρος τους από την εταιρεία αυτή. Εάν τα βουλγαρικά δικαστήρια ενεργήσουμε πραγματικά ω δικαστήρια θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική των παρόχων διότι δεν, ε, έχουν, ε, δεν έχει συνάψει η εταιρεία σύμβαση πώλησης. Υπάρχει η απόφαση C618 2010 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καθώς ε, και το άρθρο 3 του κανονισμού 805 κάθετος 2004. Παρ' όλα αυτά, οι βουλγαροί δικαστές αγνοούν τις διατάξεις αυτές. Αυτό σημαίνει κιόλα ότι ήταν ε, μάταια τα ευρωπαϊκά προγράμματα για κατάρτιση των ε, δικαστών στη Βουλγαρία. Οι δικαστές ε, λαμβάνουν οδηγίες και μεροληπτούν στις δίκες. Υπάρχουν λοιπόν εδώ σημαντικές ε, παραβιάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον δυσκολεύεται να πιστέψει ότι δεν έχουν υπογραφεί σωστές συμβάσεις. Αυτή είναι η λυπηρή πραγματικότητα που ισχύει εδώ και δεκαετίες στη Βουλγαρία. Και υπάρχουν ε, οι ε, ανώτατες ε, τιμές ενέργειας, οι οποίες επιβάλλονται όμως χωρίς καμία υπογραφή σωστής σύμβασης. Πρόκειται για παραβίαση των ε, αποφάσεων 359 11 και 411 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το να μιλά κανείς για, του, για ε, τροτούς ας πούμε ή ευάλωτους καταναλωτές ε, είναι σχεδόν ταμπού στη Βουλγαρία ο, το ανώτατο δικαστήριο τώρα ε, θα πρέπει να αποφασίσει εάν ε, θα πρέπει να εφαρμόσει τον ε, κανόνα του άρθρου 27 σχετικά με παροχή μη ετηθήσα ε, θα πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει, να λάβει άμεσα μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει αυτός ο εκβιασμός ε, και αυτές οι εκβιαστικές πληρωμές ε, που ζητάει η εταιρεία από τους καταναλωτές. Θα πρέπει να γίνει ενδεχομένως μια επίσκεψή σας επιτόπου. Εμείς έχουμε όλα τα στοιχεία της εγκληματικής διεθνείς ε, δράσεις ε, ε, ανθρώπων χωρίς καμία, κανέναν ενδιασμό που στέλνουν λογαριασμούς και παίρνουν χρήματα από ανθρώπους που δεν πρέπει να δώσουν τα χρήματα αυτά. Στην Βουλγαρία οι πολίτες είναι άνθρωποι που πρέπει να προστατεύονται. Είναι καταναλωτές ε, που πρέπει να προστατεύονται. Ε, βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 10 χρόνια ε, και πλέον και δεν είναι δυνατόν να ισχύουν τέτοιες περιπτώσεις. Στην απόφαση της υποθέσεως Σίμενταλ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βασίστηκε στην αρχή της άμεσης εφαρμοσιμότητας ενός ενωσιακού κανόνα. Εξού και όλες οι μετέπειτα εθνικές αποφάσεις οι οποίες αντιτίθενται σε αυτή την αρχή θα πρέπει να θεωρηθούν μη εφαρμοστές χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε ε, ε, να αποφασίσει επ' αυτού με τελεσίδικο τρόπο δικαστήριο εθνικό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Όσον αφορά τα ερωτήματα τα οποία έχει υποβάλει ο αναφέρον, όσον αφορά δηλαδή την ενεργειακή απόδοση και τη δημολόγηση στην ε, Βουλγαρία και όσον αφορά τα, δικαιώματα των καταναλωτών μπορώ να πω τα εξής. Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση έχει αντικαταστήσει την οδηγία για, την, ε, ε, για τις υπηρεσίες ε, ήταν πρώτερη της ενεργειακής απόδοσης και σε αυτήν την αναφερόταν αρχικά ο αναφέρον όταν έχουμε ε, πολυκατοικίες ε, οι οποίες ε, στη Βουλγαρία έχουν ένα κατακόρυφο σύστημα σωληνώσεων για τη θέρμανση, η κατάσταση όντως είναι λίγο ιδιαίτερη. Κατανοούμε ότι το συνταγματικό δικαστήριο στη Βουλγαρία έχει ε, πάρει την απόφαση ε, σε σχέση με την ε, συνδιαχείριση που έχουν αυτές οι πολυκατοικίες σε βάση του καθεστώτος συνειδιοκτησίας και αυτό δεν έχει άμεση σχέση με το ενωσιακό δίκαιο και επομένως δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε καν το θέμα της προστασίας των καταναλωτών στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά ε, τις αναφορές στο σημείο 25 της ημερησίας διατάξεως. αναφέρουμε αναφέρομαι κυρίως στην 892-2008 ε, της Μίλα Γκρέτσεβα, 1542 του κυρίου Δήμητρ Μπαλούτσεφ του 9 ε, επίσης ε, την 38 του 2013 του Ντόντσο Ντούντεβ επομένως έχουμε, ε, έχουμε αναφορές από το 8, από το 9, από το 13 και τι μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετούμε το θέμα μελετούμε το πώς έχει μεταφερθεί η οδηγία στο νομοθετικό σύστημα της Βουλγαρίας μετά μας λέει θελ ελέγχουμε εάν ε, υπάρχει παραβίαση του, ε, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σε άλλη αναφορά η Κομισιόν μας λέει ότι ο αναφέρον θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας. Αλλά τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα στην ουσία πρόκειται για αναφορές οι οποίες αφορούν το ίδιο ε, θέμα, δηλαδή το, τα δικαιώματα ε, των ε, πολιτών της Βουλγαρίας, των βουλγάρων καταναλωτών που έχουν παραβιαστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του θέματος δεν δίνει καμία απόφαση. Ε, συζητούμε, μελετούμε κτλ. Ερχόμαστε σε επαφή με τις βουλγαρικές αρχές. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει, ε, δεν έχουν τη δυνατότητα οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσουν εάν ναι ή όχι υπάρχει παραβίαση των ε, δικαιωμάτων και της προστασίας των καταναλωτών. Δεν μπορεί να απαντήσει η Κομισιόν εάν έχει παραβιαστεί επιτέλους η ενωσιακή νομοθεσία. Θα πρέπει να μας δώσει μια μια σαφή απάντηση η Κομισιόν. Γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων στο Συμβούλιο από το 2009 μέχρι το 2015. Η Κομισιόν μας λέει ότι ε, μελετά στοιχεία τα οποία κατ' εμέ είναι προφανή. Ζητώ από όλους τους παρισταμένους να μου πούν πληρώσατε τους λογαριασμούς σας θα πληρώνατε τους λογαριασμούς σας εάν δεν είχατε συμβατική ε, υποχρέωση απέναντι ε, στον πάροχο, εάν δεν είχατε σύμβαση δηλαδή με τον πάροχο ε, θα πληρώνατε τους λογαριασμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πάει στη Βουλγαρία για να δει ε, τι συμβαίνει στην ε, Σόφια. Ε, υπάρχουν γειτονιές ολόκληρες στη Σόφια που, έχουν, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό. Ζητώ επισταμένος ε, κάποιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας δώσει μια σαφή απάντηση. Όσα είδαμε μέχρι τώρα καταδεικνύουν αδυναμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ή ε, προσπάθεια αποφυγής ε, απάντησης ε, σαφούς από πλευράς της Επιτροπής. Εγώ θα ήθελα να έχω μία σαφή απάντηση στο ερώτημά του. Μου υπάρχει ναι ή όχι παραβίαση ε, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ έχουμε περίπτωση μη ύπαρξη συμβατικής υποχρέωσης. Δεν υπάρχει σύμβαση, δεν υπάρχει συμβόλαιο ε, με, ε, με τον πάροχο. Ε, εδώ δεν καταλαβαίνω τι δουλειά κάνει η Κομισιόν. Γραφειοκρατία και μόνο γραφειοκρατία χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα σαφή απάντηση. Έχουμε 10 ε, αναφορές υπό το σημείο 25 της ημερησίας διατάξεως είναι ε, αναφορές όλες αυτές που πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαλίνοφ. Νομίζω ότι πραγματικά θα συμφωνήσετε ότι δεν είναι τόσο απλό όταν υπάρχουν τόσες πολλές αναφορές ε, ε, με, τόσα, με τόσες πολλές αναφορές ε, για ένα ίδιο θέμα. Πολλές φορές ε, υπάρχουν αναφορές από πολλές χώρες που αναφέρονται στο ίδιο θέμα, αλλά τόσες πολλές για το ίδιο θέμα από μία χώρα σημαίνει ότι υπάρχουν, υπάρχει μία σειρά προβλημάτων. Άλλα που τα κληροδότησε το κομμουνιστικό σύστημα, άλλα τα οποία σχετίζονται με τεχνικές αδυναμίες, άλλα που σχετίζονται με την ανεπάρκεια των δικαστηρίων στην ε, Βουλγαρία. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, το ζήτημα το τελευταίο σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή ανεπάρκεια και μία αποτελεσματικότητα των ε, βουλγαρικών δικαστηρίων να προστατέψουν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο αναφέρον τα είπε όλα, ανέλησε πολύ καλά τα στοιχεία, αλλά το ε, ίδιο το γεγονός ότι ως ίστατη ε, καταφυγή χρησιμοποιούν οι Βούλγαροι υπήκοοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για να προσπαθήσουν να υποκινήσουν μια διαδικασία επί παραβάση σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια καλή περίπτωση να υπεραμεινθούμε της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Βουλγαρία. Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Εδώ μιλάμε όμως για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ε, που ε, επηρεάζονται αρνητικά, που προσπαθούν να διαμαρτυρηθούν στη Βουλγαρία και δεν έχουν, κάνει, δεν έχουν καταφέρει τίποτα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση το βουλγαρικό δικαστικό σύστημα δεν είναι σε θέση να δώσει απάντηση. Επομένως θα πρέπει ως ε, πραγματικά ίστατη προσφυγή να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ε, μια απάντηση έτσι ώστε ε, να καταλάβουν και οι πολίτες της Βουλγαρίας ότι η Ευρώπη είναι εδώ για να τους βοηθήσει. Επομένως, σαν επισήμως από το ΕΛΚ ζητώ να μείνει ανοιχτό το θέμα. Κύριε Κούνεβα. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή όπω ε, φαίνεται αδυνατούμε να καταλάβουμε τα προβλήματα στη Βουλγαρία και να καταλάβουμε και τη λογική των πολιτών που ζουν εκεί και αυτά που περιμένουν από εμά, προτείνω να κάνουμε μια επίσκεψη στη Βουλγαρία, να συναντήσουμε όλοι αυτοί οι οργανισμοί και πολίτε και οργανώσει και να δούμε επί τόπου τι συμβαίνει. Γιατί έχουμε αυτοκτονίες. Έχουμε πολύ σοβαρές περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με το ρεύμα, με την τέρμανση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτοί οι άνθρωποι να αυτοκτονούν και εμείς θα τους απαντάμε άλλα τα άλλα. Αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Έχουμε λίγο χρόνο. Μήπω θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει αυτά που ακούστηκαν. Σαφώς υπάρχει πρόβλημα στη Βουλγαρία. Δεν είμαι βέβαιη αν είναι πρόβλημα της ε, βουλγαρικής νομοθεσίας ή πρόβλημα της ε, μεταφοράς του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν ξέρω επίσης αν είναι πρόβλημα που συνδέεται με την κομμουνιστική κληρονομιά. Υπάρχουν ε, πολλές πολυκατοικίες όπου υπάρχουν τεχνικά προβλήματα όσον αφορά την ακριβή μέτρηση και τιμολόγηση. Έχουμε εξετάσει αναλυτικά το θέμα. Είχαμε πολλές συναντήσεις με βουλγαρικές αρχές, η τελευταία εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε τον ε, Δεκέμβριο του 2015. Επίσης είχαμε διαδικασία επιπαραβάσης στο θέμα. Θέσαμε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, σχετικά με το πώς γίνεται η τιμολόγηση. Η διαδικασία επιπαραβάση ξεκίνησε το 2012 και σύμφωνα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις και θέσαμε ερωτήσει ε, σχετικά με το εάν ε, έχει μεταφερθεί σωστά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στη Βουλγαρική Νομοθεσία. Ε, η διαδικασία μεταφοράς στο Βουλγαρικό Δίκαιο έχει ήδη κλείσει. Στη Βουλγαρική Νομοθεσία έχουν αλλάξει τα εξής. Καταρχάς, ο πρώτος κανόνας είναι ο μετρητής ε, πάντα να ε, τοποθετείται από τον καταναλωτή. Αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί για τεχνικούς λόγους. Έτσι επιτρέπει η τιμολόγηση να γίνεται ανάλογα με την κατανάλωση. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την οδηγία που προβλέπει στο άρθρο 93 ο μετρητής ε, για την θέρμαση να τοποθετείται εφόσον ε, αυτό είναι εφικτό από τεχνικής πλευράς ε, και αποδοτικό όσον αφορά το κόστος και το όφελος. Ακριβείς μετρητές λέει θα πρέπει να τοποθετούνται όπου αυτό είναι αποδοτικό όσον αφορά την ισορροπία κόστους όφελους. Και σε περιπτώσεις όπου είναι δυνατή τοποθέτηση τέτοιων οικονομικών μετρητών ε, για τις οριζόντιες εσωληνώσεις και για ε, ξεχωριστά κτίρια. Το θέμα είναι πώς υπολογίζονται οι λογαριασμοί για διαμερίσματα. Το αποτέλεσμα της σχετικής έρευνας έδειξε ότι το κόστος είναι σχετικά χαμηλό για κάτι τέτοιο. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι το κόστος ε, είναι πάνω από αυτό που προβλέπει η οδηγία. Επίσης υπήρξαν διάφορες ερωτήσεις ε, σχετικά με τη μεθοδολογία για, την, ε, για τον καταμερισμό του κόστους θέρμανσης. Στο άρθρο 93 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση υπάρχει επιπλέον διάταξη που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να υιοθετούν διαφανείς κανόνες όσον αφορά τον καταμερισμό του κόστους. Μέρος αυτών των διαφανών κανόνων ε, συνδέεται με το κόστος τοποθέτησης, ε, μάλλον το κόστος της εγκατάστασης ε, στο κτίριο. αν ο καταναλωτής θέλει να διακόψει την παροχή θέρμανσης προς το διαμέρισμά του, θα πρέπει να πληρώσει για να γίνει σχετική εγκατάσταση στο κτίριο. γεγονός ε, λοιπόν ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ε, λόγω ενεργειακής ένδυας έχουν ε, διακόψει την παροχή θέρμασης προς το διαμέρισμά τους. Παρόλα αυτά σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν για την εγκατάσταση του κτηρίου. Για συνταξιούχους και χαμηλόμισθους αυτό μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους ο ενεργειακός λογαριασμός. Αλλά το άρθρο 9.3 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση προβλέπει να υπάρξει τέτοια δυνατότητα και επίσης το ε, Συνταγματικό Δικαστήριο έχει εξετάσει το θέμα αυτό και εξέτασε τις ε, σχέσεις ε, με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των υπηκών της Βουλγαρίας. Εξετάσαμε την περίπτωση για να δούμε μήπως υπάρχει παραβίαση του ε, ε, ενωσιακού δικαίου. Δεν διαπιστώσαμε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Η σύμβαση ανάμεσα ε, στην Ένωση Ιδιοκτητών και τον επιμέρους ιδιοκτήτη βρήκε το Σταγματικό Δικαστήριο ότι είναι νόμιμη. Στη Βουλγαρία υπάρχουν νόμοι κοινωνικής προστασίας. Και έτσι μπορούν να ζητήσουν ε, επιδοτήσεις οι Βούλγαροι υπήκοοι. Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν ελλείψεις ε, στο νόμο αυτό. και το πρόβλημα συνεχίζει να είναι άκρος προβληματικό. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι το θέμα των δικαιωμάτων ιδιοκτησία ε, συνεχίζει να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επίσης, όσον αφορά τις δικαστικές πρακτικές των δικαστηρίων της Βουλγαρίας, και το θέμα εάν ε, μεμονωμένος διοκτήτης μπορεί να σταματήσει την παροχή ενέργειας προς το διαμέρισμά του. σε σχέση και με την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Ε, υπήρξε ε, αίτημα του διαμεσολαβητή προς το ανώτατο δικαστήριο να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ποιο πρότυπο πρέπει να ισχύει. Αν θα πρέπει δηλαδή εδώ να υπερισχύει η οδηγία για την προστασία του καταναλωτή ή η ενεργειακή νομοθεσία. Ο χρόνος που χρειάζεται ένα βουλγαρικό δικαστήριο δεν είναι υπερβολικός. Ελπίζω λοιπόν αυτό κάπως να απαντάει στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο το θέμα αυτό, το οποίο επηρεάζει πολλούς πολίτες μας. Όπως πολύ σωστά υπόθηκε, η Επιτροπή Αναφορών ε, είναι το τελευταίο μέρος όπου μπορούν να προσφύγουν ε, οι πολίτες και ε, δεν μπορούμε να μην ακούσουμε αυτά που μας λένε οι πολίτες. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους Ευρωβουλευτές ε, ακούσαμε αντίθετες ε, απόψεις. Προτείνω η Επιτροπή Αναφορών να έρθει σε επαφή με τις βουλγαρικές αρχές και να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Στο μεταξύ, θα ήθελα να συστήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξάγει περαιτέρω έρευνες με βάση αυτά που υπόθηκαν σήμερα. Είμαι βέβαιη ότι Αυτά που ακούσαμε από τους ευρωβουλευτές ε, είναι έγκυρες πληροφορίες και γνωρίζουν τι λένε. Ε, νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ερευνήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό, να αφήσουμε ανοιχτή ε, την αναφορά αυτή και ως Επιτροπή Αναφορών να στείλουμε επιστολή στις βουλγαρικές αρχές για να διαπιστώσουμε εμείς οι ίδιοι πώς έχει η κατάσταση για να μπορέσουμε κιόλας ε, να λάβουμε πιο εμπεριστατωμένη απόφαση. Προτείνω λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή. Η κυρία Κούνεβα θα ήθελε το λόγο, παρακαλώ. Συγχωρείτε ε, να διευκρινίσω κάτι να έχουν υπόψη όταν μελετάνε και όταν συζητάνε με, τις, ε, με τους εκπρόσωπους ε, των κυβερνησιών. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πώς λειτουργεί η Βουλγαρία και τι συμβαίνει εκεί. Σε ένα άλλο θέμα. Είναι ε, τώρα η κρίση στην Ευρώπη και θα πάρα πολλοί Βούλγαροι στη Βουλγαρία και χάνουν τις δουλειές τους στις χώρες που ζούσαν μέχρι τώρα. Και πάνε να γραφτούν στο ΟΑΕΤ να δηλώσουν ότι είναι άνεργοι. Και τι συμβαίνει. Του λένε ναι καλά, αλλά τώρα το σύστημα είναι μπλοκαρισμένο. Δεν μπορείτε να γραφτείτε. Ελάτε κάποια άλλη μέρα. Φεύγουνε, πάνε άλλη μέρα. Έτσι, πολλές φορές δεν μπορεί να γραφτεί ο πολίτης ότι είναι άνεργος. Κάποιοι που του έχει πάρει το πείσμα, κάθονται και λένε εγώ θα περιμένω μέχρι να ανοίξει το σύστημα σήμερα γιατί δεν το καταφέρνω άλλη, άλλη μέρα να έρθω και έτσι γράφονται. Και αυτή τη στατιστική με αυτόν τον τρόπο που παίρνουμε δηλώνεται πώ έχει μειωθεί η ανεργία στη Βουλγαρία. Έχουν βρει κόλπα, έχουν βρει μετόντου που να παρουσιάζουν τα πράγματα πολύ καλά, νόμιμα, κανονικά και το υπόβατρο να είναι χάλια. Αυτό είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κούνεβα που μας δίνετε περισσότερες πληροφορίες για το τι συμβαίνει. Ωραία. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της εξέτασης αυτών των αναφορών. Όπως είπα προηγουμένως, θα μείνουν ανοιχτές μέχρι περαιτέρω διερεύνησή τους. Μάλιστα. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 28. αναφορές από επικόους Μαλτέζικης και Βρετανικής Ιθαγένειας. Δεν είναι εδώ οι αναφέροντες. Με ενημερώνουν όμως ότι έχει υπάρξει ενημέρωση που σας έχει μοιραστεί κιόλας. Αν δεν κάνω λάθος. Οι αναφορές 1737 του 2013, 341 του 2014, 1655 του 2014, 2102 του 2014 και 24 του 2015. Δεν παρίστανται οι αναφέροντες. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν γέννη, η Μαλτέζικη νομοθεσία προβλέπει διαφορετικές χρεώσεις για την ηλεκτρική ενέργεια και το νερό με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Επομένω. Οι κάτοικοι και μη κάτοικοι λαμβάνουν διαφορετικές χρεώσεις λοιπόν. Ε, και αυτή η διαφοροποίηση των τιμών ε, οδήγησε στην υποβολή επιμέρους αναφορών. Οι αναφορές έχουν θίξει επιμέρους ε, ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν ε, να τα πάρουμε τη σειρά, ε, αν με επιτρέπετε. Έχουμε τρία διαφορετικά ζητήματα, ουσιαστικά. Το πρώτο είναι η πρόσβαση στο μειωμένο τιμολόγιο γενικά για τους υπηκόους. Την 2102 και την 24-2015. Το δεύτερο είναι η πρόσβαση ε, των κατοίκων για την ε, μείωση τα μειωμένα τιμολόγια 1655-2014, 341-2014. Και το τρίτο ζήτημα είναι η πρόσβαση των ε, κατοίκων σε πληροφορίες ως προς την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που αφορά την 341-2014. Όπως είπα λοιπόν, η νομοθεσία ε, στη Μάλτα προσβλέπει διαφορετικές χρεώσεις. Ε, επομένως, για να καταφέρουν οι πολίτες να λάβουν αυτό το μειωμένο τιμολόγιο, πρέπει ε, να, υπάρξει, να υπάρξουν αντίστοιχες πληροφορίες από την εταιρεία τιμολόγησης. Εν γέννη, οι Ευρωπαίοι πολίτες βλέπουν ότι η εταιρεία αυτή έχει ζητήσει συγκεκριμένε ε, διοικητικέ διαδικασίες για να δώσει τις ε, πληροφορίε προκειμένου να ενταχθούν στο μειωμένο τιμολόγιο. Υπήρξε επαφή με τις μαρτεζικέ αρχές από το 2011, ε, δεν ήταν ικανοποιητική απάντηση, ξεκίνησε η διαδικασία επί παραβάση, μετά οι αρχέ στη Μάλτα άλλαξαν την τακτική του. Σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτε δικαιούνται να κάνουν αίτηση στην εταιρεία Unlimited απλώς κάνοντας μία αίτηση μαζί με την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους. Επομένως έχει λυθεί αυτό το ζήτημα, είναι σαφές. Στη συνέχεια, οι Μαλτέζικες αρχές οδήγησαν, ε, δημιούργησαν και μία ε, διαδικασία δικαστική, ας πούμε, ειδική για όσους ήθελαν να αποζημιωθούν και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η διαδικασία λειτουργεί καλά. Επομένως, έχει ληφθεί για τις δύο από τις αναφορές το κύριο ζήτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους, ε, τη 1655, για παράδειγμα, οι αναφέροντες ενημέρωσαν ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα για να ενταχθούν στο μειωμένο τιμολόγιο. Οι Ευρωπαίοι πολίτε αυτοί ή γενικά άτομα που θέλουν να ενταχθούν στο τιμολόγιο πρέπει να κάνουν αίτηση με την υπογραφή του ιδιοκτήτη, αν ήταν ενοικιαστέ οι ίδιοι. Έπρεπε λοιπόν να λάβουν και τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη για να ενταχθούν στο μειωμένο τιμολόγιο. Η Επιτροπή είχε έρθει σε επαφή το 2014 με τις Μαλτέζικε Αρχές. Το Μάιο του 2016 οι αρχέ της Μάλτας ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι θα αλλάξουν την πρακτική τους και θα επιτρέπουν στους ενοικιαστέ ε, να εποφελούνται των μειωμένων τιμών και χρεώσεων χωρί τη συνένεση του ιδιοκτήτη. Θα πρέπει μόνο να υποβάλουν αντίγραφο ε, της συμφωνίας μίσθωσης. Συμφωνεί η Επιτροπή. Ε, βρισκόμαστε ακόμα σε επαφή με τις αρχές της Μάλτας για αυτό το ζήτημα. Απλώς ε, είναι για να διευκρινίσουμε ε, ίσονα, ζητήματα. Όμως η γενική προσέγγιση είναι σωστή πλέον. Για αυτές τις τέσσερις τώρα αναφορές και το γενικό ζήτημα της διαφοροποίησης τιμών, ο Εμμανουέλ Βάλετς, ο συναδελφός μου, θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγορά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να προσθέσω ε, ορισμένες πληροφορίες που συνδέονται με το θέμα της διάκρισης μεταξύ καταναλωτών ε, βάσει του τόπου ε, διαμονής τους, κατοικίας τους. Σε ό,τι αφορά τον, την κατηγορία υπηρεσιών, εμπίπτει στα πεδία εφαρμογή του άρθρου 20 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες της Εσωτερικής Αγοράς του 2006, που απαγορεύει ε, τη διάκριση στην αντιμετώπιση ε, των καταναλωτών με βάση τον τόπο κατοικίας τους, εκτός και αν αυτό ε, αιτιολογείται από αντικειμενικά κριτήρια. Η αιτιολογική σκέψη 95 της οδηγίας αυτής υπενθυμίζει τις επιμέρους κατηγορίες αντικειμενικών κριτηρίων που θα μπορούσαν ενδεχομένω να επικληθούν οι, οι εμπορευόμενοι για να ε, παράσχουν τις υπηρεσίες τους και να κάνουν αυτή τη διάκριση στις τιμές πιο συγκεκριμένα. Εν προκειμένου, είναι αρκετά δύσκολο από τη δική μας κοπιά να δούμε ποια μπορεί να είναι εδώ τα αντικειμενικά κριτήρια που να αιτιολογούν αυτή τη διάκριση στη μεταχείριση. Βλέπουμε ότι οι μη κάτοικοι συστηματικά ε, παρεμποδίζονται από το να επωφεληθούν πιο ευνοϊκών ε, ε, χρεώσεων σε σχέση με τους κατοίκους, που είναι πιο εύκολο για αυτούς δηλαδή να, να πάρουν αυτές τις μειωμένες τιμές. Και βλέπουμε κάτι στο φάκελο που να αιτιολογεί αυτή τη διακριτική μεταχείριση. Ιδίω ό,τι αφορά το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια και την παροχή του, ένα στοιχείο που ενδεχομένω θα μπορούσε κανεί να επικληθεί ε, είναι το γεγονό ότι οι κάτοικοι αυτοί πληρώνουν τους φόρους τους στην ε, χώρα προέλευσής τους. Όμως, εδώ να υπενθυμίσω ότι το δικαστήριο έχει αποφανθεί ρητός ότι Ε, μπορεί να θεωρηθεί ε, το φορολογικό καθεστώ ω αντικειμενικό κριτήριο, όμω θα πρέπει να υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του φόρου που έχει επιβληθεί και ε, τη εφαρμογή αυτού του προνομιακού καθεστώτο τιμών. Και δεν βλέπουμε εδώ ποια είναι αυτή η άμεση σύνδεση μεταξύ των δύο. Επίσης διαπιστώνουμε ότι οι Μαλτέζικες Αρχές έχουν ανακοινώσει τη δημοσιοποίηση κατευθυντηρίων γραμμών guidance δηλαδή, για τους παρόχους υπηρεσιών για το άρθρο 9α ε, στην ε, οδηγία για τις υπηρεσίες στην εστρική αγορά. Το άρθρο 20 όντως έχει μεταφερθεί ε, στις Μαλτέζικες, ε, στη Μαλτέζικη νομοθεσία με το αντίστοιχο άρθρο 9α. Υπάρχει λοιπόν διάταξη τέτοια και στο Μαλτέζικο Δίκαιο που να απαγορεύει την διακριτική μεταχείριση. Ως εκ τούτου, εμείς δεν έχουμε λάβει γνώση της επίσημης δημοσιοποίησης αυτής της κατευθυντηρίας γραμμής. Όμως, ε, από ό,τι βλέπουμε, κινούνται προς σωστή κατεύθυνση και οι καταναλωτές μπορούν να βασίζονται σε αυτές τις κατευθύνες γραμμές για να ε, ζητούν την διόρθωση αυτής της κατάστασης από τις αρμόδιες αρχές. Κλείνοντας, Να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Μαΐου ε, υπέβαλε πρόταση κανονισμού για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς το ζήτημα αυτό της διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Ε, ένα σχέδιο κανονισμού που δημιουργεί συγκεκριμένα δικαιώματα εφαρμοστέα ακριβώς για αυτούς τους καταναλωτές με σκοπό να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτές τις καταστάσεις. Μελετούμε την κατάσταση τη στιγμή για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε ε, ιδίω για, την, για τη Μάλτα. Όμω και πάλι το σχέδιο κανονισμού έχει στόχο ακριβώ να απαντήσει σε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Με ενημερώνουν ότι υπάρχει τρίτος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλετε να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, Θα ήθελα να αναφερθώ στο συγκεκριμένο θέμα της πρόσβασης στα δεδομένα κατανάλωσης. Αυτό σχετίζεται με την αναφορά 341, όπου ε, ισχυρίζεται ότι ως ε, ενοικιαστής ε, δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωσης, ε, μόνο ο ιδιοκτήτης έχει. Σύμφωνα με τη δική μας εκτίμηση, είναι απολύτως ε, νόμιμο να έχει τη σύμβαση με την εταιρεία παροχής ε, ενέργειας ο ιδιοκτήτης ε, ακόμα και όταν έχει ενοικιαστεί το διαμέρισμα. Ωστόσο, ο ενοικιαστής θεωρείται ο τελικός πελάτης, ο τελικός καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και αν είναι κανεί ενοικιαστή, ε, επιτρέπεται πρέπει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωσή του, ακόμα και αν, έχει... ακόμα και αν δεν έχει υπογράψει ο ίδιος τη σύμβαση με τον ε, πάροχο. Τούτου λεχθέντος, Η νομοθεσία έχει εφαρμοστεί σωστά στο Μαλτέζικο δίκαιο και σύμφωνα με την νομοθεσία ο ενοικιαστής έχει πρόσβαση στα δεδομένα εφόσον τα ζητήσει. Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι ο αναφέρον ζήτησε τα δεδομένα αυτά. Ούτε ήρθε σε επαφέ με το μηχανισμό επίλυσης διαφορών που έχουν θεσπίσει οι αρχές της Μάλτας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο αναφέρον έχει δίκιο ότι πρέπει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωσή του, ωστόσο δεν βλέπουμε να, έχουμε, να έχει αναλάβει τα απαραίτητα βήματα για να πετύχει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει εδώ εκπρόσωπος των αρχών τη Μάλτας που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλου. Θα ήθελα Καταρχάς, να επισημάνω ότι τα θέματα που θίγονται σε αυτές τις αναφορές και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προέρχονται, δεν, δεν είναι θέματα νομοθεσίας. Η εθνική νομοθεσία δεν κάνει διακρίσεις με βάση την υπηκότητα. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπήρξαν περιπτώσεις όπου η πρακτική εφαρμογή του νόμου έχει οδηγήσει σε προβλήματα όσον αφορά την, ε, την παροχή ενέργειας σε τιμές κατοίκων της Μάλτας ε, καθώς και στην ε, πρόσβαση των δεδομένων κατανάλωσης, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλλον θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναγνωρίζει τη δουλειά μας και που θίγει το θέμα της ε, παράβασης όσον αφορά τις τιμές για κατοίκους. Προτείνουμε λοιπόν κλείσιμο των αναφορών ε, στα θέματα αυτά. Στο άλλο θέμα που σχετίζεται με την σχέση ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, όπως είπαν ήδη οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε αναλάβει βήματα για να ε, αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αλλάξει τις διοικητικές πρακτικές στο θέμα αυτό. Και έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης ε, τη σχέση αυτής ε, και χωρί την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ώστε ο ενοικιαστή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωση. Θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία για να τονίσω ότι το θέμα ιδιοκτητών ε, ενοικιαστών δεν έχει να κάνει μόνο με μη κατοίκου με μη υπηκόους της Μάλτας, να... είναι θέμα που αφορά και υπηκόου τη Μάλτας. Δεν είναι λοιπόν θέμα που σχετίζεται με την υπηκότητα. Το προσώπου. Um, um, στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναγνωρίζει τη δουλειά που έχουμε κάνει και στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να κλείσει και αυτή η αναφορά προς όφελος και των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέκερ θα ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να επικροτήσω την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξει διευκρίνηση και ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την ε, σύναψη ενεργειακών συμβάσεων ε, για κατοικίες. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες ε, και είναι από τα πράγματα που περιμένουν οι πολίτες από την Ευρώπη. Να αποφύγουμε δηλαδή τις περιπτώσεις που έχουν οδηγήσει σε σύγχυση σε κράτη-μέλη. Μήπως μπορείτε σύντομα να μας πείτε πότε αναμένεται η σχετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει στον κύριο Μπέκερ. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτά. Το ερώτημα αφορά το περιεχόμενο της νομοθετικής προτάσεως που σχετίζεται με την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης και αν κατάλαβα καλά και του γεωαποκλεισμού. για αυτό το θέμα, σε σχέση με το σημερινό μας ζήτημα, οι διατάξεις είναι αρκετά απλές. Η πρόταση κανονισμού απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση που βασίζεται άμεσα ή έμεσα στην εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής. Όταν και εφόσον η υπηρεσία παρέχεται στον τόπο εγκατάστασης ε, του ε, παρόχου ε, της υπηρεσίας ή στον τόπο που έχει επιλέξει ο πάροχος της υπηρεσίας. Όταν ε, μιλάμε για παροχή επομένως υπηρεσίας επιτόπου, ε, είτε πρόκειται για ενοικίαση αυτοκινήτου, είτε πρόκειται για ξενοδοχειακή μονάδα, είτε για παροχή νερού ή ηλεκτρικού και από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαφορά εφαρμοστέου δικαίου, δεν υπάρχουν αντικειμενικά πιο σημαντικά κόστη για την παροχή ε, μιας υπηρεσίας η διαφορά της φορολογίας δεν υφίσταται, διαφορά δυσκολίας ή βαθμού δυσκολίας δεν υφίσταται και επομένως δεν μπορεί να δικαιολογηθεί διαφορετικό κόστος. Ε, τα αντικειμενικά κριτήρια λοιπόν ε, δεν ε, υπάρχουν και μόνο βάσει διαφορετικών κριτηρίων αντικειμενικών μπορεί κανείς να αιτιολογήσει διαφορετική τιμολόγηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε την πρόταση στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και ε, η συγκήτρια η κυρία Ρόζα Τούνα. Αυτά μπορώ να σας πω σχετικά με το κείμενο αυτό. Ο κύριος Πέκερ και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Η ερώτησή μου όμως είχε να κάνει με το ότι είπατε ότι τον Μάιο συμφωνήσατε να προτείνετε ρύθμιση και θα ήθελα και η συγκεκριμένη μου ερώτηση ήταν πότε θα δούμε την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Η απάντηση είναι δύσκολη θα εξαρτηθούν όλα από την εξέλιξη της νομοθετικής διαδικασίας. Δεν μπορώ να σας πω. Δεν είναι πλέον το θέμα αυτό στα χέρια της ε, Κομισιόν. Η Κομισιόν έκανε ε, την ε, πρόταση, την υπέβαλε την 25η Μαΐου. Άρχισε άμεσα και γρήγορα η εργασία στο Συμβούλιο και δυστυχώς δεν μπορώ να προβλέψω κάτι διαφορετικό. Παρακαλώ πολύ, κύριο Γιάρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν συμβαίνει πάντα να... Υπάρχει εκπρόσωπος ε, της ε, Κομισιόν. Δεν συμβαίνει όμως πάντα να έχουμε εκπρόσωπο της ε, εμπλεκόμενης χώρας. Ε, χαίρομαι λοιπόν για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια έκκληση προς τη Γραμματεία. Συχνά έχουμε αναφορές όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχει ε, παραβίαση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς ή ότι υπάρχουν διακρίσεις. Θυμάμαι για παράδειγμα μια περίπτωση για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων. και τη διαφορά των ε, τιμών. Άλλη περίπτωση που θυμάμαι ήταν η χρήση γης όπου υπήρχε διάκριση για ανθρώπους μιας ηλικίας και πάνω. Βλέπω λοιπόν ότι η Κομισιόν ε, αρχίζει να ασχολείται με τέτοια θέματα, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πού επιτρέπεται λοιπόν τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν μόνα τους ε, και πού έχουμε περιπτώσεις διακρίσεων. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε σχετική διευκρίνηση. Και όσο πιο προσεκτικά εξετάζουμε το θέμα, τόσο πιο δύσκολα είναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χαίρομαι που ακούμε μια θετική απάντηση. Η Κομισιόν λέει ότι ναι, εντάξει, είναι κάπως προβληματική υπόθεση, αλλά και το ε, ε, εμπλεκόμενο κράτος μέλος λέει ότι ναι, υπάρχουν όντως κάποια προβλήματα τα οποία ε, μπορούν να διορθωθούν. Θα ήθελα λοιπόν ε, και στις ε, περιπτώσεις ε, που σας ανέφερα πριν να έχουμε σχετική διευκρίνηση. Άλλωστε ο συνάδελφος Μπέκερ έχει μια ηλικία. Νομίζω ότι θεωρείτε και εσείς κάπως ε, ε, ε, προβληματικές της διακρίσεις λόγω ηλικίας και ένας ηλικιωμένος μπορεί να είναι γεωργός. Εν αυτό είναι άλλη ιστορία. Πάντως, χαίρομαι για τη συζήτηση και για τις θετικές παρεμβάσεις που, ακούσαμε. Μπράβο, έρχεται. I'm wondering Αναρωτιέμαι μήπως ε, οι, εκπρόσωποι της Μαλτέζικης κυβέρνησης ε, θέλουν να απαντήσουν. Όχι από ό,τι φαίνεται. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε ποια από αυτές ε, τις αναφορές έχουν ε, έχουν αντιμετωπιστεί ήδη και ποιες προτίθεστε να αντιμετωπίσετε ε, στο εγγύς μέλλον. Έχετε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Ποιες αναφορές λοιπόν ήδη έχουν αντιμετωπιστεί. Η Κομισιόν νομίζω σε ορισμένα σημεία ήταν πάρα πολύ σαφής ενώ σε άλλα λιγότερο σαφής. Πριν πάρουμε απόφαση θα ήθελα ε, να δώσω την ευκαιρία στους εκπροσώπους της κυβέρνηση της Μάλτας να αποσαφηνίσουν τα πράγματα. Okay, and so... Λοιπόν, κοιτάξτε, οι αναφορές οι οποίες σχετίζονται με την ε, παραβίαση την οποία ε, ανέφεραν ε, οι εκπρόσωποι της Κομισιόν. Ήταν σαφής η Κομισιόν στην προσέγγιση της. Και επιβεβαιώνουμε λοιπόν ότι αυτές έχουν αντιμετωπιστεί οι αναφορές. αυτές μπορούν να κλείσουν γιατί έχουμε ανταποκριθεί ε, και έχουμε ανταποκριθεί λοιπόν στις διοικητικές ε, ε, στις διοικητικές διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει πριν μερικούς μήνες. Μπορείτε να μας πείτε όμως, λέει πρώτα συγκεκριμένα ποιες αναφορές είναι. 21.02 του 2014 αυτή η αναφορά και 0024 του 2015. They specifically deal λέτε ότι αυτές είναι οι συγκεκριμένες αναφορές που αφορούν διαδικασία παραβάση. Μπορεί να επιβεβαιώσει η Κομισιόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει διαδικασία παραβάση και θεωρεί η Κομισιόν, μπορεί να μας το πει συγκεκριμένα, ότι δεν, δεν υπάρχει πρόβλημα απέναντι των αρχών. Απάντηση της Κομισιόν, ναι, τα θέματα τα οποία αφορούσαν διαδικασίες επί παραβάση από πλευράς της Κομισιόν ε, έχουν λήξει. Να προτείνω λοιπόν αυτές οι συγκεκριμένες αναφορές να κλείσουν, 2102 και 0024. Φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποια εκκρεμή ζητήματα με τις άλλες αναφορές για τις οποίες χρειαζόμαστε και περισσότερες πληροφορίες και σαφέστερη απάντηση από την Κομισιόν από ό,τι καταλαβαίνω και από την Κομισιόν και από τις αρχές της Μάλτας θα μας δοθούν ε, όσον ούπο αυτές ε, οι επιπλέον ε, πληροφορίες. Επομένως αφήνουμε ανοιχτές τις τρεις πρώτες αναφορές και κλείνουμε την 2102 και τη 0024. Συμφωνείτε πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η εργασία μας σήμερα το πρωί. Πολύ ωραία τα είπαμε, πολύ χρήσιμα ήταν όλα αυτά που ακούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ε, αναφέροντες ε, που ε, ήρθαν, που μας άκουσαν, που μας έστειλαν το βίντεο. Ευχαριστούμε τις αρχές που παρίσταντο. Καλές διακοπές.